καταλογίζει και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Και κατόπιν ε, της αναδείξεως της κυρίας Νταντσίλα ως Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, επίσης ε, διαπιστώνουμε την χειρία της έδρας της από 21 πρώτο 18. Επίσης ε, γνωστοποιήθηκε ότι την κυρία Νταντσίλα θα αντικαταστήσει η κυρία Γκαμπριέλα Ζωάνα. Καλώς όρισε, συνάδελφος, η οποία θα είναι τακτικό μέλος του Κοινοβουλίου και θα έχει ε, πλήρες αρμοδιότητες και δικαιώματα όπως προβλέπει ο κανονισμός. Η νομική